Uh, Καλησπέρα σε όλους σας. Αρχίζει η συνεδρίαση της Επιτροπής τώρα και θα το γυρίσω στα Σουηδικά. Eh, λοιπόν, σας καλωσορίζω και στα Σουηδικά όλους ε, στην Επιτροπή. Μετά τις ελληνές διακοπές αρχίζει και πάλι η δουλειά και συγκεκριμένα με ψηφοφορίες σήμερα. Αλλά να, να πάμε με τη σειρά. Πρώτον, συνεδρίαση των συντονιστών. Δεύτερον, έγκριση της ημερήσιας διάταξης χωρίς αλλαγές. Θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σημείο 3. Και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι ε, θα έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 9 Οκτωβρίου. Στις 9 Οκτωβρίου λοιπόν ο ειδικό εισηγητής ε, των Ηνωμένων Εθνών θα παρευρεθεί ε, ειδικό συγητής για θέματα βίας κατά των γυναικών. Αλλά όλα αυτά θα τα κοινοποιήσουμε. Ε, ξανά σε όλους σας. Τέσσερα, ανακοίνωση του Πρόεδρου σχετικά με τις στάσεις των συντονιστών. Στα έγγραφά σας έχετε τα πρακτικά. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας προτείνω εγώ, να προσθέσω τίποτα και θεωρώ ότι εγκρίνουμε και τα πρακτικά αυτά που ήταν το σημείο 5. Έγκριση των πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων 13-14 Ιουλίου του 2011 και 29 και 30 Αυγούστου του 2011 πάλι. Εάν δεν διαφωνεί κανείς, θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά. Και περνούμε μέσω στις ψηφοφορίες. δημιουργία χρηματοδοτικού μέσου για την αναπτυξιακή συνεργασία. Η κυρία Κράτσα είναι η συγγήτρια. Έχει το λόγο. Παρακαλώ κυρία Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω να συμπληρώσω ιδιαίτερα πράγματα από αυτά που είπαμε την τελευταία φορά όταν εξετάσαμε τις τροπολογίες. Ήθελα να ευχαριστήσω τις συναδέλφους που στο, γενικά στο, σε, σε κοινό πνεύμα προσέθεσαν διαστάσεις που εμπλούτησαν τη γνωμοδότησή μας. Πιστεύω ότι γίνεται σαφές ότι απαιτούμε αφενός η γυναικεία διάσταση να ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας και αφετέρου ότι τονίζουμε ότι χρειάζονται ξεχωριστά χρηματοδοτικά μέσα διότι χρίζουν ε, <clears throat> χρήζουν ακόμη ανάγκης ε, οι γυναίκες παντού ειδική παρέμβασης για την άρση των διακρίσεων και για τη δημιουργία συνθήκων ένταξης στην οικονομική ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κράτσα. Αρχίζουμε λοιπόν. Στα αγγλικά θα κάνω τις ψηφοφορίες όπως συνηθίζω. Συμβιβαστική 4. Ψήφι υπέρ τη συμβαστική. 4 κατά άποχε, εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική υπαριθμό 5 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν Συνεπώ πολλέ τροπολογίε και φτάνουμε στην 9. Η τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, ζητώ συγγνώμη, ξέχασα να θέσω σε ψηφοφορία την τροπολογία 46. Ακριβώς πριν την 9 θα πρέπει να ψηφίσουμε τη 46 πρώτα. Ψηφί υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη 49 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 50 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 καταπίπτει, η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωρούμε στην 51 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η 56 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 13, η τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα θα πάμε στην 59, προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς να εξετάσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Όχι. Θα την ψηφίσουμε τότε. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχο. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 60 παρακαλώ. Εγκρίνεται. Η 15 ψηφί Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Άρα η 16 καταπίπτει. Η συμβαστική 8 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 67 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα η 19 καταπίπτει. Ψηφίζουμε την 20. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 κατά πίπτη. Ψηφίζουμε την 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχο. 78. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά λοιπόν την 78. voting Μου έκλεψαν την ε, κάρτα ψηφοφορία μου, λέει η κυρία Κονέλη. Βασικά το πορτοφόλι ήθελα, αλλά μαζί με το πορτοφόλι μου πήραν και την κάρτα. 79. Υπέρ. Κατά απόχέ. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά απόχέ. Νομίζω ότι χρειάζεται έλεγχο και η 80. Παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφτεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ή 87 υπέρ. «87 παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται». Η 88 υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω χρειάζεται έλεγχο η 88. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Απορρίπτεται. Η 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ερχόμαστε στην τροπολογία 28, 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα οι 2 κατά πίπτη. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 34 τώρα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 5 καταπίπτει και ψηφίζουμε την 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα το σύνολο του ψηφίσματος ηλεκτρονικά παρακαλώ αρχίζει τώρα η ψηφοφορία And the is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σαφέστατα. Ευχαριστώ πολύ ε, την κυρία Κράτα. We then continue to... Συνεχίζουμε Ψηφίζουμε για τον προϋπολογισμό. Η κυρία Χάνι είναι εδώ, δεν θα πάρει το λόγο προφανώς. Ξεκινούμε την ψηφοφορία. 62 τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. να ξαναρχίσουμε νομίζω. Να το ελέγξουμε. Ελέγχουμε 62-21. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62 0-0. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62-23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62-03. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 62-03. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62-04. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. 62-04. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62-17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62-05. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 6206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6222 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62.07 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62.08 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62.09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6210 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6224 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62-18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62-12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62-30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6-2-19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6-2-13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6-2-14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6-2-15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 2 13 υπερ κατα αποχες εγκρινεται 6 2 14 υπερ κατα αποχες εγκρινεται 6 2 15 υπερ κατα αποχες απορριπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο. Όχι, δεν ψηφίζουμε το σύνολο. Αστιεύομαι. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ψηφίζουμε λοιπόν για την ε, έκθεση για το 2011 για την ε, ε, συνεργασία των πολιτικών για την ανάπτυξη. Να δώσω το λόγο στην κυρία Τσέσκοβα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις αυτές. Θα ήθελα να πω ότι με έκπληξή μου είδα ότι κάποια σημεία τελικά θα μείνουν εκτός κειμένου. Αυτό φάνηκε μετά την ψήφιση των τροπολογιών. Όμως τον Ιούλιο όταν συνεδριάσαμε στην Επιτροπή μας, δεν συνεδριάσαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί είχαμε πολλές απουσίες και τότε δεν ε, προβλήθηκαν καθόλου αντιρρήσεις για τα σημεία αυτά. Και μάλιστα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής επισήμαναν ότι η έκθεση που εγώ έχω συντάξει είναι αποδεκτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία σας και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ε, ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα σχόλια. Προχωρούμε λοιπόν ε, στην ε, ψήφιση του σχεδίου γνωμοδότησης. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οι 3 και οι 5 καταπίπτουν. Ψηφίζουμε όμως την 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 και 10 είναι ταυτόσιμες ποιος είναι υπέρ τις 9 και τις 10 διανατάσσεως χειρός κατά αποχές εγκρίνονται 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Για την 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25. Ψηφίζουμε την 25. ή να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 24. Καλώς. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την τροπολογία υπαριθμών 24. Πέρας. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 και 28. Είναι ταυτόσιμες τροπολογίες και συμβατές ως προσθήκη στην τροπολογία 25. Ψηφίζουμε την 26 και την 28. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 26 και την 28. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 29 αποσύρεται. Ψηφίζουμε την 27 λοιπόν. Θα ψηφίσουμε την 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορώ να καταλάβω να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για την 32 έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 33. Ποιος είναι υπέρ της 33. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δυσκολεύομαι να καταλάβω. Ε, να το ελέγξουμε, να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 33. Πέρας. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αυτό σημαίνει ότι θα ψηφίσουμε την 35 και την 38, οι οποίες είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ αυτών των δύο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 36. Ψηφίζουμε την 36. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37 λοιπόν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 εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Okej, okay, då eh, går jag tillbaks till att eh, prata svenska. Λοιπόν, επιστρέφω στα σοϊδικά, αν επιτρέπετε. Αφού έληξε η ψηφοφορία μπορώ να συνεχίσω να μιλώ τη μετρική μου γλώσσα. Πάμε στο επόμενο σημείο της μισής διατάξης. Σημείο 9, ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη του Φόρου Επιρρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ιστότητα των Φύλων, του Φόρουμ EIGE, e, συνοπτικά. Η πρώτη, μάλλον σήμερα θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, με τα μέλη της Επιτροπής μας. Αυτή τη στιγμή συστάθηκε α, αυτό το φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να ακούσουμε εμπειρίες. Είναι εξαιρετική λοιπόν αυτή η ευκαιρία που μας δίνεται. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας για αυτή τη συζήτηση, οπότε δεν θέλω να καταγραφώ πρώτο του χρόνου για να σας παρουσιάσω ξεχωριστά. Σας καλωσορίζω θερμά την κυρία Μαντράγκα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 Ευχαριστώ πολύ, επαναλαμβάνω, για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Για λόγους χρονικούς ε, δεν θα συστηθώ. Πριν από τρία χρόνια σας είχα εκτενώς ε, παρουσιάσει ε, το ιστορικό μου και πώς ασχολούμαι θέματα διακρίσεων και επελέξετε και μεταξύ άλλων υποψηφίων να με διορίσετε σε αυτό το φόρουμ εμπειρογνωμόνων και νομίζω αυτό αρκεί ως εισαγωγή. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα και αυτό που μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι γίνεται με το φόρουμ αυτό, πώς πάει. Και καλά και άσχημα. Τι εννοώ. Να πούμε πρώτα τα καλά. Μετά τα λιγότερο καλά. Στη συνέχεια θα σας αναφέρω δύο λόγια για το δικό μου και το δικό μας ρόλο για ενδεχομένω ε, πιθανές βελτιώσεις και θα κλείσω με μία έκκληση που θα ήθελα να σας απευθυνώ να σκεφτείτε πάρα πολύ καλά το μέλλον. Τα καλά. Σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση στο Ινστιτούτο. Αρχίζει να καταρτίζει και να καταθέτει εκθέσεις Έχουμε ένα κέντρο τεκμηρίωσης για συγκεκριμένα θέματα όπως είναι για παράδειγμα η βία κατά των γυναικών. Ε, γίνεται κατάρτιση, εκπαίδευση και ε, δικτύωση για διάφορα θέματα. Και το Σαββατοκύριακο θα ε, λάβετε και το newsletter μας με πάρα πολλές εκθέσεις και δραστηριότητες και πεπραγμένα. Και σας λέγω επίσης ότι ήρθε και η ώρα για αποτελέσματα. Βεβαίω, παρακαλώ και την επίκειά σα, Είναι πολύ δύσκολο από το τίποτα να στήσει κανείς ένα τέτοιο Ινστιτούτο να προσελκύσει προσωπικό, να κάνει έρευνες και αυτό χρειάστηκαν ε, μερικά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. Ε, κοστίζει και πολύ χρόνο. Ε, ευτυχώς έχει έρθει η ώρα τώρα να δρέψουμε τους καρπούς των προσπαθειών μας. Και δεν θα σας μιλήσω για την ουσία των εκθέσεων και το τι αναφέρετε, που θα μπορούσατε να αποκομίσετε μόνοι σας ε, ε, άποψη. Τώρα έρχομαι στα ζητήματα που πηγαίνουν λιγότερο καλά, τα άσχημα και εκείνα που χωλένουν. Κατά την άποψή μου να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτό το λέει και η νομοθεσία, και για τη διοίκησή μας και για το δίκτυο εμπειρογνωμόνων ε, έχει κάποιες αρμοδιότητες. Εντάξει, μπράβο της και πολύ καλά και συμφωνώ, αλλά ε, το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό ε, όπου διεξάγονται όλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει υψηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο διεύθυνσης δηλαδή και διοίκησης και στο φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Το είπα και στην Βελίντα Μπάικ ε, εκείνο τον καιρό, αλλά δυστυχώ ήταν άκαρπη αυτή η προσπάθεια. Τώρα για το προσωπικό και τη διοίκηση ε, του Ινστιτούτου μας. Εγώ είμαι Ολλανδέζα και έχω συνηθίσει να λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια και θα το κάνω. Αν κοιτάξει κανείς απ' έξω το προσωπικό, διαπιστώνει δύο πράγματα. Έχουμε πάρα ε, πολλούς συνεργάτες, υπαλλήλου που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα ε, ως προς την ισότητα των φύλων, ε, των ευκαιριών, τη διαφοροποίηση. Μπορεί να έχουν σπουδάσει γυναικεία θέματα, θέματα φίλου και σίγουρα ο καθένας είναι ειδικό στο θέμα του, στατιστικολόγος, τεκμηριωτής, αλλά σε ό,τι αφορά το φίλο, πολλές φορές αυτά είναι θεωρητικά από τα βιβλία. Πολλοί δεν έχουν ζήσει στο πετσί τους, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει να είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας και να σου φέρονται έτσι. Και όταν έχεις ένα τέτοιο Ινστιτούτο σαν το δικό μα, θα πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστή. Να είναι υπάλληλοι ε, γνώστες του θέματος, να ξέρουν ποια είναι η κακία που <laughs> τους περιβάλλει. Και κατά την άποψή μου δεν είναι δεδομένο αυτό. Και κάτι άλλο που επίσης είναι ανεπαρκές είναι η γνώση της πολιτικής από πλευράς υπαλλήλων. Διαπίστωσα ότι διάφοροι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν καν πώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. άκουσαν άκουσα Διαφορά ανάμεσα στα θεσμικά όργανα Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινοβούλιο. Ε, μέχρι ένα επίπεδο μπορεί κάπω να τον ντύσει αυτό τεχνικά, αλλά από πολιτική άποψη να ξέρει πώ δουλεύουν τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, α πούμε, ότι ο κύριο Ολάντ είναι το υπαριθμό ένα πρόσωπο στην ε, Γαλλία. Έχει σημασία ε, ποιος επίτροπος και από ποιο πολιτικό κόμμα προέρχεται. Ε, τι επιρροές ε, έχει στην εργασία στη χύψη χώρα των γυναικών ε, η τραπεζική κρίση έχει σημασία. Όταν ακούω ότι γίνονται σκέψεις για διαπραγμάτευση και πάλι των κριτηρίων της πλατφόρμας του Πεκίνου ε, και τι αυτό θα μπορούσε να αποδώσει. Ανησυχώ και λέω κοιτάξτε προσοχή πώς έχει σήμερα η πολιτική κατάσταση. Πολλοί από τους υπαλλήλους δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει καθημερινά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ε, γίνεται στη δική σας Επιτροπή, στην ημερήσια διάταξή σας. Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο γίνονται εκθέσει, λαμβάνουν χώρα κάποιε δραστηριότητε που δεν έχουν πραγματική σύνδεση με την καθημερινή πολιτική. Συστάσει απευθύνονται όσο και καλά τεκμεριωμένε να είναι επιστημονικά αυτές, λαμβάνουν πολύ ε, λίγο υπόψη τους την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα, πραγματικά, αμαρτία. Και πίσω τύπος αδιαφορεί. Όπως βλέπετε, το ξέρετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, προσελκύσει κανείς το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων για θέματα φύλου. Και πάλι αυτό δεν έχει να κάνει με την καθημερινότητα, γιατί δεν είναι κάτι που θα συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, οπότε ο τύπος αδιαφορεί. Οπότε κάνουμε διάφορες δραστηριότητε και ασκήσεις, ε, άχρηστες. Στο φόρουμ εμπειρογνωμών ακούω πάντα από το διευθυντή ότι ε, ναι, αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε και το πρόγραμμα εργασίας που έχουμε. Εντάξει, να λειτουργούν οι υπηρεσίες, αλλά και σε ένα πρόγραμμα εργασίας να υπάρχει αρκετός χώρος ε, να αντιμετωπίζεται και η επικαιρότητα. Α είναι. Σας είπα ότι το δίκτυο εμπειρογνωμόνων και η δίκτυα στον πληθυντικό αρχίζουν να λειτουργούν ε, και είναι γεγονός. Πολλοί εμπειρογνώμονες συμμετέχουν από πολλά κράτη-μέλη. Αυτό όμω όλα αποδίδουν. Ειλικρινά δεν ξέρω. Ελπίζω να λειτουργεί αυτό το Ινστιτούτο. Αλλά οι εμπειρογνώμονες με τους οποίους συζητώ λέγουν όλοι ε, ανεξαιρέτως ότι δεν ξέρουν αν το μήνυμά τους περνάει και δεν ξέρουν τι γίνεται με τη δική τους πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή αυτοί τα λένε, αλλά ε, ε, δεν είναι μεγάλη η σύνδεση του Ινστιτούτου με τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε ε, τώρα στο δικό μου ρόλο ή το δικό μας ρόλο. 18 εκπρόσωποι είναι η διοίκηση και στο φόρουμ των εμπειρογνωμόνων εκπροσωπούνται τα κράτη-μέλη αλλά και συχνά υπάλληλοι, εμπειρογνώμονες ε, πολλές φορές ε, από την ε, επιστήμη και ανεξάρτητοι όπως εγώ και εργοδότες, συνδικάτα, λόμπι γυναικών, επιχειρηματίες, γυναίκες κτλ. Δύο είναι οι μεγάλες ομάδες εργασίας πλέον. Το ένα έχει να κάνει με τους δείκτες του Πεκίνου και το άλλο ε, με το δίκτυ φίλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω την τιμή να, ε, να προεδρεύω στη δεύτερη ομάδα εργασίας. Και στην ομάδα, στο φόρουμ Εμπειρογνωμών ε, και στις ομάδες εργασίας έχουμε το ίδιο πρόβλημα, αυτό που σας είπα για το δίκτυο. Γίνονται προτάσεις, ε, αλλά δεν ξέρουμε τι αποτέλεσμα έχει αυτό και αυτό αποθαρρύνει, απογοητεύει. Μέχρι τώρα ήταν πολλοί εκείνοι που έδιναν στο Ινστιτούτο ελαφρυντικά ε, και κάποια περίοδο χάριτος, αλλά τώρα έχει, αρχίσει, έχει έρθει η ώρα της αλλαγής φρουράς. Ε, και σου λένε οι ότι φτάνει πια. Εγώ α, έχω άλλα πράγματα να κάνω καλύτερα. Δεν μπορώ να χάνω το χρόνο μου εκεί αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ανησυχητική εξέλιξη και ελπίζω ε, η διοίκηση ε, του Ινστιτούτου να αντιδράσει γρήγορα. Βεβαίως είναι δύσκολο να λειτουργεί μια τέτοια δομή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διοίκηση, Εμπειρογνώμονες, Φόρουμ και Κόντρα Φόρουμ. Ε, τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά μας όμως. Και όπως γνωρίζετε, εσείς έχετε διορίσει δύο εμπειρογνώμονες. Δύο αναπληρωτές. Μάλλον, ε, εγώ είμαι το τακτικό μέλος και η Ισπανίδα συνάδελφος είναι αναπληρώτρη. Ε, αλλά πάντα κάποιος εκπροσωπεί την Επιτροπή σας εκεί. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε εμείς και μόνο εκ του λόγου του γεγονότος ότι καμιά φορά οι εκπρόσωποι των κρατών μελών εκεί δεν τολμούν να κάνουν προτάσεις. Διότι φοβούνται Πώς χάσουν το κεφάλι τους. Εμείς δεν φοβόμαστε τον αποκεφαλισμό, έπρεπε να σα πω. Αλλά δεν έχει νόημα να πηγαίνουμε εκεί μόνο να καθόμαστε και να μην ανταλλάσσουμε με εσά απόψε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην αρχή, μετά ε, από κάθε συνεδρίαση έστελνα στη γραμματεία σας εδώ μια έκθεση αλλά άκουσα ότι δεν, δεν τη στέλναν στους βουλευτές αυτή την έκθεση. Εκεί σταμάτησα κι εγώ να γράφω εκθέσεις. Ε, ε, βέβαια αυτό μπορεί να μην είναι κάτι που με τιμά, αλλά κι εγώ άνθρωπος είμαι. Καλό θα ήταν να στέλνετε και ένα μέλος της γραμματείας στο φόρουμ και να σημειώνει ε, αυτά που συζητούμε εκεί και να σας τα διαβεβάσει το κάνατε και θα θέλαμε να μας είχατε ενημερώσει κύριε Πρόεδρε εκ των προτέρων ότι θα γίνει αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω. Η επικοινωνία δεν πάει καλά. Ε, πριν το καλοκαίρι η κυρία Λάγκμπακ ήρθε εδώ η διευθύντρια του Ινστιτούτου. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας είχατε καλέσει και εμάς. Δημόσια συνεδρίαση είναι, το ξέρω, αλλά δεν βλέπω κανένα εδώ από τη διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και κανονικά θα πρέπει να τους ενδιαφέρει αυτά που έχουμε να σας πούμε, να τα ακούσουν γιατί τους αφορά. Εάν ανανεώσετε το διορισμό μου και ελπίζω να το κάνετε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε πώς θα επικοινωνούμε. Παράδειγμα, κάποιος από εμά να έρχεται δυο φορές το χρόνο, τουλάχιστον στους συντονιστές οπωσδήποτε και να σας ενημερώνει, αλλά να ενημερώνετε και από εσά. Και τέλος, να πω και κάτι για τη Βιέννη. Υπάρχει μια φήμη επίμονη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει, λέει, να ε, συγχωνεύσει το ΆΕΚΕ και ε, το Φόρουμ για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Ε, αυτή η φήμη επιμένει πάρα πολύ, δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Θα πρέπει να διευκρινιστούν τα πράγματα το συντομότερο και καλό θα ήταν να το συζητήσετε κι εσείς και να ξέρετε τι γίνεται. Ένα Ινστιτούτο για το φύλλο. Τι νόημα έχει και τι κέρδος ε, θα έχει αν συγχωνευτεί με το Ινστιτούτο της Βιέννης. Σε θέματα ρατσισμού και εθνοτήτων, τι σχέση έχει αυτό με το φύλλο. Μέχρι τώρα αυτό το Ινστιτούτο για το ρατσισμό αποδείχθηκε ότι ήταν Ινστιτούτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν ε, αφορά μόνο το ρατσισμό και τις ε, διακρίσεις με βάση την εθνικότητα. Νομίζω ότι σας τα είπα έτσι τα σίκα σίκα και τις κάφη Σταματώ εδώ και περιμένω με μεγάλη χαρά τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Καλησπέρα σας σε όλες και όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είμαι κάπως άρρωστη. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι προσυπογράφω απόλυτα τα λόγια της ε, συναδέλφου Βίλιαμ. Δεν θέλω να επαναλάβω λοιπόν και εγώ τα ίδια όσα ήδη εκείνη ε, σας επικοινώνησε να πω ότι συμμερίζομαι πλήρως από τα λεγόμενα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι εγώ Ορίστηκα ως πρώτο πνευματικό μέλος ε, στο φόρουμ των εμπειρογνωμόνων και για λόγους που δεν μπορούσα εγώ να επηρεάσω, κατάφερα να είμαι παρούσα στις 6 από τις 9 ε, συνεδριάσεις του φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα, ταυτόχρονα όμως που δημιούργησε μια κάποια ανασφάλεια, γιατί ποτέ δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη για την συνέχεια των εργασιών, ώστε να μπορέσω και εγώ να αφοσιωθώ στην ολοκλήρωση κάποιων ε, τέτοιων εργασιών, όπως η Πιούλη ε, που είναι το τακτικό μέλος, ε, συμμετείχε σε όλες τις εργασίες και εγώ πραγματικά ένιωθα ένα παράπονο γιατί δεν μπόρεσα να συμμετάσχω σε κάποιες συνεδριάσεις και δεν ήξερα ακριβώ ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχή ε, που μου αναλογούσε στον πληρωματικό μέλο. Με το πέρας του χρόνου κατάλαβα ότι η συμμετοχή δική μου ουσιαστικά ήταν ταυτόσιμη με αυτή του τακτικού μέλους. Οι συμμετοχές μου λοιπόν σε αυτές τις συνεδριάσεις ήταν πραγματικά ο χρόνος και ο τόπος που ρίχναμε να έχουμε μια ανταλλαγή ουσιαστικών απόψεων και για διάφορα θέματα βεβαίως. προσπαθώντας και εγώ να σταθμίσω τα υπέρ και τα κατά του Ινστιτούτου και του Φόρουμ, ναι, αυτό μπορώ να πω και εγώ, είναι ότι χρειάζεται πιο πολλούς χρόνος, χρειαζόταν πιο πολλούς χρόνος για να ζητώ θέματα. Ήτανε μάλλον συνεδριάσεις εξπρέστα, έλεγα, με κλειστή ημερήσια διάταξη, και ήταν δύσκολο πραγματικά να στήσουμε σε βάθος πολλά ζητήματα. Εκεί εκπροσωπούνται φορείς διαφόρων φορέων και χωρών και κάποιες ε, φορές δίνεται δυνατότητα να ακούγονται απόψεις και φωνές από όλους τους φορείς ε, και τα κράτη-μέλη σχετικά με το πώς βλέπουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι το θετικό. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή εγώ ποτέ δεν ήμουν σίγουρη κατά πόσον θα μπορώ να συμμετάσχω στην επόμενη συνεδρίαση ή όχι, καθώς ήμουν αναπληρώτρια, αυτό οδηγούσε μια μηχανία, γιατί κάθε φορά έβλεπα καινούργια πρόσωπα και όταν βλέπεις συνέχεια καινούργια πρόσωπα είναι δύσκολο να πεις ότι παρακολουθείς τις εργασίες ε, ολοκληρωτικά και όχι κατακαιρματισμένα. Τέλος πάντων, έτσι είχαν τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά το φόρμα, τα τελευταία τρία χρόνια, είδαμε ότι το, Ινστιτούτο, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων μεγαλώνει. Μεγαλώνει και αλλάζει, αλλάζει το προσωπικό του μπαίνουν νέοι άνθρωποι με μεγάλη διάθεση για εργασία και με όραμα και όπως ε, μιλούσατε και εσείς πριν λίγο τον προπολογισμό και αυτό είναι ένα θέμα αγώνα και μάχης πολύ συχνά και για το Ινστιτούτο, ένα Ινστιτούτο που μάχεται για την ισότητα και εμείς στο φόρουμ των εμπειρογνωμόνων ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά για μας να ανταλλάσσουμε απόψεις για αυτά τα ζητήματα και ήταν πολύ καλό πραγματικά γίνεται αυτή η αλλαγή απόψεων ε, καθώς εκπροσωπούνταν τόσοι φορείς. Το να ξεκινά από το μηδέν ένας νέος φορέας, ε, ξέρετε, είναι κάτι πολύ δύσκολο, ιδίω όταν εκπροσωπεί έναν ε, μεγάλο οργανισμό όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν αυτό γίνεται μέσα από μία μικρή και περιφερειακή, αν θέλετε, χώρα της Ευρωπαϊκής όπως είναι η Λιθουανία. Και αυτό πρέπει να το προσμετρήσουμε, πιστεύω, στα θετικά. Παρά τα αυτά, αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι όλο το έργο που έχει γίνει αυτά τα τελευταία χρόνια από το Ινστιτούτο δεν έχει ε, την αναγνώριση που του αναλογεί, διότι εδώ και χρόνια γίνεται δουλειά κατάρτιση και καλύτερη οργάνωση του οργανισμού και είναι ένας οργανισμός, ένα Ινστιτούτο, άγνωστο στην Ευρώπη τελικά, και όταν μιλάμε για έναν οργανισμό που μάχεται υπέρ της ισότητας. Κάποιες φορές έχω την αίσθηση ότι δεν του δίνεται η πρωταγωνιστική θέση που το αναλογεί. Και δυστυχώς δεν αποτελεί και σημείο αναφορά στην Ευρώπη όπως θα έπρεπε. Γιατί το λέω. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις, τουλάχιστον η δική μου άποψη είναι, ή όπως είπε και Γουέλιν. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε μεταξύ άλλων στο φόρουμ είναι στο μέτρο του δυνατού πρώτα απ' όλα να διαφημίσουμε την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Αυτού Ινστιτούτου και δεύτερον να διαδώσουμε, να διαφημίσουμε το έργο που κάνει. Σε αυτή μας την προσπάθεια λοιπόν τότε συνειδητοποιήσαμε πόσο άγνωστη είναι η ίδια η ύπαρξη και το έργο αυτού του Ινστιτούτου. Κάτι λοιπόν που μου τράξει την προσοχή, δεν ξέρω αν είναι σωστό να το πω, αλλά θα ήθελα να το πω γιατί μου τράβηξε την προσοχή. Το έργο που γίνεται από αυτό το Ινστιτούτο, από τις γυναίκες που έχουν συνέλθει σε αυτό το Ινστιτούτο και προσπαθούν, θεωρώ ότι είναι τεράστιο αναλογικά με τη διαφήμιση και την προβολή που δεν του δίνεται. Άρα λοιπόν η διάδοση και η προβολή του έργου είναι πολύ σημαντική για να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ισχύ και δύναμη και να αποτελούν σημείο αναφορά τέτοιοι φορεί. Ξέρετε, και πριν από τρία χρόνια θυμάμαι ότι εδώ προτείναμε ένα είδος οδικού χάρτη, αν θέλετε, για αυτό το Ινστιτούτο και εγώ είχα πει ότι καλύτερο να μιλήσουμε για πιο συγκεκριμένε δράσεις, για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και γρήγοροι στις ε, κινήσεις μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά εγώ αυτό που ήθελα της εξ αρχής είναι συγκεκριμένες δράσεις από τον Ινστιτούτο. ώστε να αποτελεί το σημείο αναφοράς στα κράτη-μέλη και στους αρμόδιους φορείς ισότητας των κρατών μελών. Εννοείται ότι τον πρώτο ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τον εκτελεστικό ρόλο σε αυτά τα προγράμματα, ναι, αλλά και μέσω λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να ε, μεταλαμπαδευτούν και να εφαρμοστούν αυτά τα προγράμματα ε, στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς όμως αυτό δεν έγινε πράξη. Θέλω να πω ότι η στρατηγική επικοινωνία ε, όπως έγινε αφορά και πριν, η στρατηγική λοιπόν επικοινωνίας ήταν καλυμμένη. Ακούστηκαν πολλά στρατηγική επικοινωνία ώστε να γνωστοποιηθεί το έργο του Ινστιτούτου. Πιστεύω λοιπόν στρατική ήταν καλή, αλλά ίσως για οικονομικούς λόγους ή γιατί είναι δύσκολο να φτάσει αυτό το έργο με τον κατάλληλο τρόπο σε 27 κρατη Τελικά θα πρέπει να γίνει πιο πολλή δουλειά, πιο πολλή προσπάθεια στον τομέα της επικοινωνίας μέσα των κοινωνικών δικτύων. Λοιπόν, έχουμε δουλειά να κάνουμε μπροστά μας, ώστε να γνωστοποιήσουμε καλύτερα αυτό το έργο. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να γνωστοποιηθεί και ο διαγωνισμός που γίνεται και κάθε χρόνο έχουμε και το ετήσιο ημερολόγιο για τις γυναίκες που εμπνέουν την Ευρώπη. Λοιπόν, γίνονται τέτοιες προσπάθειες επικοινωνίας, αλλά δεν αρκούν. Γιατί δεν είναι πράξεις που αρκούν για να γνωστοποιήσουν επαρκώς το έργο του Ινστιτούτου, Κάτι γνώμη μου. Η αδυναμία που μπορούμε να εντοπίσουμε, τουλάχιστον εγώ εντοπίζω, σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο, είναι ότι είναι άγνωστος οργανισμός και δεν αποτελεί σημείο αναφορά στην Ευρώπη. Και ξέρετε και κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι ότι αν αυτό το Ινστιτούτο έδινε υποτροφίες ή επιχορηγήσεις, αυτό θα ήταν ένα άλλο μέσο για να προβληθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι δυνατό από πλευράς οικονομικών πόρων της Ένωσης, αλλά τέτοιου είδους υποτροφίες και επιχορηγήσεις θα βοηθούσαν το έργο και την προβολή του Ινστιτούτου. Τώρα για το μέλλον. Το μέλλον του Ινστιτούτου. Μετά από πέντε χρόνια από την σύσταση του Ινστιτούτου, από την αρχική συμφωνία για τη σύστασή του, πιστεύω ότι μετά από πέντε χρόνια είναι καιρός να λανσάρουμε ξανά αυτό το Ινστιτούτο. Δηλαδή έχουν περάσει πέντε χρόνια με ομάδες εργασίας, με τα στοιχεία, με ε, σχέδια επιχάρτου. Καιρός να περάσουμε στην πράξη. Μπορεί αυτά που λέω να είναι δύσκολα, αλλά εν τέλει για να μπορέσει να εκτιμήσει, κανεί, να κανείς τη σημασία ενός τούτου είναι βλέποντας τις πράξεις, τις δράσεις του. Δράσεις που θα φέρουν εις πέρα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχουν θετηθεί για το επόμενο διάστημα. Σε θέματα λοιπόν ισότητας ε, στις ε, απολαβές, στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αύξηση των γυναικών στις θέσεις λήψης αποφάσεων, αυτή είναι το μυς που από κοινού με, την, το κόσμο μπορούν να γίνουν πολλά με την ευελιξία στο ωράριο εργασίας και την προσπάθεια συμφιλίωσης του εργασιακού με τον οικογενειακό βίο τι είναι τομεί όπου μπορούμε πραγματικά να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι σημαντική τομή για τι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση σαν γέννη. Καλό επίση θα ήταν να γίνει παράλληλα και κάτι για την βία με γνώμονα το φύλλο, δράσεις που μπορούν να ξεκινήσουν από το ίδιο Ινστιτούτο και να υλοποιηθούν στα κράτη-μέλη. Επίσης, ο ρόλος των ανδρών εν προκειμένου στη νέα κοινωνία, τη νέα ισότιμη κοινωνία που επιζητούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλουμε δηλαδή το Ινστιτούτο να επεξεργαστεί στρατηγικές και να δείξει το δρόμο στα κράτη-μέλη όλοι δουλεύουμε, ίσως με διαφορετικούς ρυθμούς και με διαφορετικό τρόπο, αλλά όλοι επεξεργαζόμαστε αυτά τα ζητήματα, όλοι μας απασχολούν. Καλό λοιπόν να έχουμε κοινέ στρατηγικέ. Είναι θέματα δική σημασία για το μέλλον όλων μα, ώστε να μπορούμε να μιλούμε για μια Ευρώπη που χαρίζεται από την ισονομία όλων των πολιτών. Αν Επίσης, επιβάλλουμε και κυρώσεις στα κράτη-μέλη για τη μη τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για θέματα γεωργικής, πολιτικής, μεταφορών περιβάλλοντος. Αν λοιπόν γίνεται αυτό, θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχουν κυρώσεις για μη την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για θέματα ισότητας των φύλων. Και επίσης σε επίπεδο ε, φόρουμ μερογνωμόνων ε, ε, διευθυντικού συμβουλίου, όπως και σε εθνικό περιφερειακό ή άλλο επίπεδο φορείς που δουλεύουν στο θέμα της ισότητας των φύλων θα πρέπει να ενισχυθούν όλοι αυτοί οι φορείς. Κλείνοντας θέλω να πω ότι διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς όπως είναι η δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γυναικών όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό να δώσετε κατάλληλα εργαλεία και μέσα στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για να μπορέσει να φέρει σφαίρες αποτελεσματικά το έργο Αυτά α, εν αναμονή των ερωτήσεών σας είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τις δύο ομιλήτριες. Μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ για το ανοιχτό σας πνεύμα και για την μεγάλη σας ειλικρίνεια. Είχαμε μια πολύ ανοιχτή επικοινωνία μόλις τώρα και αυτό είναι πολύ καλό πιστεύω. Μας ταιριάζει, είναι κάτι που επιθυμούμε και είναι πολύ καλό το γεγονός που ήρθατε. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στους υπολείπους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κυρία Μπάουερ παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την ειλικρίνειά σας και για τις απόψεις σας. Ανησυχώ κι εγώ για... και στεναχωριέμαι που δεν παρευρίσκεται η διοίκηση ε, του Ινστιτούτου. Τους καλέσαμε. Ήταν δυστοκία Προφανώς η δημιουργία του Ινστιτούτου αυτό είναι γεγονό, το βλέπουμε κι εμείς. Και ακούμε τι λέτε κι εσείς. Ότι δεν είναι σημείο αναφοράς για κανέναν άλλον. Παρόλο που την ίδια στιγμή ιδρύθηκαν και τα δύο Ινστιτούτα και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για θέματα φύλων και το ε, άλλο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Βιέννης από ό,τι φαίνεται δεν έχει βρει το δρόμο του ε, για να παίξει το ρόλο που του αναλογεί αυτό το Ινστιτούτο. Θα πρέπει να γίνει σημείο και πόλος αναφοράς για τους υπολείπους. Ε, είδαμε ότι διοργανώνεται διάφορα εργαστήρια, βγάζετε και ημερολόγια, πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι να κάνετε τέτοιες δραστηριότητες μόνο. Το πρόβλημα, το βασικό μέλημά σας θα πρέπει να είναι αλλού. Και πολύ συχνά έχουμε την αίσθηση κι εμείς ότι είναι συγκεκριμένη η κατεύθυνση που ακολουθεί το Ινστιτούτο. Υποστηρικτική προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Αυτό δεν είναι από μόνο αρνητικό, αλλά δεν είναι βασικός ε, λόγος ύπαρξης και δημιουργίας ε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Δεν έχει ούτε πραγματική έδρα, ούτε το απαραίτητο προσωπικό. Ε, δεν μπορούμε πέντε χρόνια να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Και κάτι άλλο που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι ότι Ο στόχος δεν είναι να ασχολούμαστε μόνο εμείς με την πολιτική του φίλου ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να το υλοποιούμε ε, το εκάστοτε πρόγραμμα, αλλά να γίνει το Ινστιτούτο αυτό ανεξάρτητο όργανο και να αναπτύσσει έργο και δραστηριότητες εποφελής για όλους. Έχετε δίκιο για την επικοινωνία. Δεν είναι ιδεώδεις οι σχέσεις και οι επαφές όχι μόνο μεταξύ της διοίκησης και του φόρουμ, αλλά πιθανότατα και μεταξύ ε, του Ινστιτούτου ΕΓΕ και του, και του Κοινοβουλίου του ίδιου. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ ε, ανησυχητικό για μας. Είπατε ότι διαπιστώνεται μία τάση και κυκλοφορούν φήμες ε, για συγχώνευση του Ινστιτούτου των Φίλων με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Βιέννης. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας θεωρούμε ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει πολύ ευρύτερο ορίζοντα και πολύ μεγαλύτερο πεδίο ε, δραστηριοτήτων και ευθύνης. και δεν μπορεί να ασχολείται με όλα. Δηλαδή σε αυτά τα θέματα φύλου δεν μπορεί παρά επιφανειακά να τα εξετάζει μόνο επιπόλαια ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και εκεί καλείται το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να εμβαθύνει και να τα μελετά σε βάθος και να ελέγχει που βρίσκονται τα προβλήματα. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα της ε, ουσίας ε, του αντικειμένου με το οποίο θα επιφορτίζεται το Ινστιτούτο. Εμείς όταν κάνουμε μελέτες στο Κοινοβούλιο, πολλές φορές τις αναθέτουμε σε εξωτερικούς. Ε, με αποτελέσματα πολλές φορές φρικτά. Πριν από δύο χρόνια ζητήσαμε μια μελέτη για την άδεια μητρότητας και πήραμε κάποιες μελέτες που ήταν πολύ κακής ποιότητας. Ανεπίτρεπτη ήταν αυτή η έκθεση. Για αυτά τα θέματα δεν είναι ε, όμως στιγμιαία. Ε, είναι θέματα που μας απασχολούν πάγια και οι μελέτες και η πραγματογνωμοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται στο πόδι. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Γιατί δεν μπορούμε να ζητούμε αυτέ τι μελέτες από το Ινστιτούτο αυτό, εξάρτητες και να το αναθέτουμε σε τρίτους ε, που είναι αμφιβόλου ποιότητα. Και αυτό δεν είναι θέμα του ΦΡΑ, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ε, ξεπερνάει το πλαίσιο του. Και σε ό,τι αφορά τώρα την απαλλαγή για το 2010, εγκρίθηκε μια πρόταση να συγχωνευθούν οι δύο οργανισμοί, αλλά δεν ξέρω από ποιον προήλθε η πρόταση. Δεν ήταν δική μας Επιτροπής Γυναικών, αλλά εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. Και αυτό οφείλουμε να το σημειώνουμε. Μπορεί εμεί να διαφωνούμε στην Επιτροπή ε, Ισότητας των Φύλων, να έχουμε πιο στεναρή άποψη. Αλλά το ζήτημα αυτό τη συγχώνευση ε, θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας όσο δεν υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στην ιστοσελίδα σας εσείς αναφέρετε απτά χειροπιαστά αποτελέσματα. Το τελευταίο διάστημα βλέπω περισσότερες πληροφορίες από ό,τι στο παρελθόν, αλλά έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι η ευκαιρία που έχουμε σήμερα με τη δική σας παρουσία εδώ μπορεί ή θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί καλύτερα. Και όταν έλθει προς συζήτηση ετήσια έκθεση, τότε θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε και τα δικά σας ζητήματα. Εμείς δεν έχουμε ιδέα ποια θέματα σας απασχολούν και τι διαπραγματεύεστε. Εκεί δεν μπορούμε και κάθε μήνα να συζητούμε αυτό το, θέμα, αλλά κάθε εξάμεινο και όταν έρχεται η συζήτηση της ετήσιας έκθεσης, μία φορά και μία δεύτερη στη συζήτηση για τον προπολογισμό αλλά να κοιτάμε και θέματα ουσίας. Και να ακούμε και εσάς, όχι μόνο το Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και για την ειλικρίνειά σας. Και ελπίζω να ε, προχωρήσουμε Και αν εμείς ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα, και να μην υποστηρίζονται αυτέ οι απόψει στο Κοινοβούλιο ότι δεν χρειαζόμαστε αυτού του οργανισμού, είναι πανάκριβοι, δεν κάνουν δουλειά, τι νόημα έχουν. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα για να μπορούμε να σα υπερπιστούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις δύο εμπειρογνώμονες, διότι μας παρουσίασαν πολύ έγκυρα στοιχεία, αλλά και διότι επέδειξαν το θάρρος και την ειλικρίνεια να επισημάνουν τα προβλήματα έτσι ακριβώς όπως έχουν. Και θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε η κυρία Μπάουερ, ότι πρέπει να εμβαθύνουμε στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν εμάς, στην Επιτροπή μας για τα θέματα των γυναικών, αλλά θέλω και να σχολιάσω κάποια θέματα που έχετε θέσει εσείς. Στους κόλπους της δικής μας Επιτροπής, το θέμα της βελτίωσης της επικοινωνίας μεταξύ ισότητας και επικοινωνίας μένει έκρεμες, έκρημη, έκρεμη, καθώς και το θέμα του πώς θα παρακολουθούνται οι φάκελοι και πώς θα μοιράζονται τα στοιχεία και τα δεδομένα εκατέρωθεν. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας σε δύο πράγματα. Πρώτον, ορατότητα. Δεύτερον, χρησιμότητα. Η αξιοπιστία όλων μας εξαρτάται από αυτές τις δύο λέξεις κλειδιά. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν την ορατότητα των δράσεών μας. Πιστεύω ότι χρειάζεται να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να έχουμε πιο απτά πράγματα να δείξουμε. Ερωτώ, λοιπόν την πρώτη ομιλήτρια. Είπατε ότι ε, προσφέρουμε τη συνεισφορά μας, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει με αυτή Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε αυτό, πώς θα γίνουν πιο αξιοποιήσιμα τα στοιχεία του Ινστιτούτου. Καλό είναι να έχουμε αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία, αλλά δεν θα πρέπει να μην μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη και τα οποία ουσιαστικά το μόνο που θα κάνουν είναι να συνεχίσουν να ε, τροφοδοτούν ε, τη φήμη που κυκλοφορεί υπέρ της συγχώνευσης αυτών των δύο ιδρυμάτων. Και δεν είναι φήμη, προβάλλονται και επιχειρήματα πολύ σημαντικά και μάλιστα σε καιρού οικονομικής κρίσης τα επιχειρήματα αυτών που θέλουν τη συγχώνευση αυτών των δύο ιδρυμάτων ε, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Ε, ευτυχώς όμως έχουμε πολύ πιο ισχυρές ε, αντιδράσεις από πλευράς Ινστιτούτου ω προς αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί υπογραμμίσατε τα κενά και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Θέσατε το θέμα του επίπεδου των εμπειρογνωμόνων. Εξεπλάγει. Το ομολογώ. Ε, ε, το, για το ότι υπάρχουν εμπειρογνώμονες που δεν είναι καλά καταρτισμένοι, που δεν γνωρίζουν τα πρακτικά ζητήματα ή τη διάσταση του φύλου στο σύνολό της. Ρωτώ λοιπόν, τι προτείνετε εσείς για την επιλογή των καταλήλων ανθρώπων με την επαρκή κατάρτιση, ποια πρέπει να είναι τα κριτήρια επιλογής και πώς θα διασφαλίζεται η διαφάνεια, ώστε ε, να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι οι εμπειρογνώμονες που δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά τα θέματα πράγματι ανταποκρίνονται σε σαφώς προκαθορισμένα κριτήρια. Από εκεί και πέρα θέλω να επανέλθω στο, θέμα της στρατηγικής. Χαίρομαι διότι βλέπω ότι το Ινστιτούτο για το 2013 θα εφαρμόσει μια πολύ συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση και με τα εθνικά σημεία επαφής. Ερωτώ όμως ε, πώς θα, πώς σκέφτεστε ότι θα βελτιωθεί αυτή, αυτό το μοίρασμα των πληροφοριών μεταξύ της δικής μας Επιτροπής για τις Γυναίκες και του Ινστιτούτου. Πώς θα βελτιώσετε την ορατότητα ε, των εργασιών του Ινστιτούτου. Πώς ε, πιστεύετε ότι μπορεί το Ινστιτούτο να παρακολουθήσει ε, τις εργασίες της Επιτροπής μας. Υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός που έχετε και πώς ε, μπορείτε να συνεισφέρετε στα θέματα που αποτελούν ε, τον καθημερινό μας κύκλο εργασιών, αν θέλετε. Όλα αυτά θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνεργασία μας. Γνωρίζετε ότι στη δική μας Επιτροπή, στο Ευρωκοινοβούλιο, οργανώνουμε δημόσιες ακροάσεις για να εξετάσουμε βαθύτερα συγκεκριμένα θέματα και πολύ συχνά απουσιάζει το Ινστιτούτο στις δημόσιες ακροάσεις μας αν σκεφτούμε τις δύο-τρεις τελευταίες που έχουμε οργανώσει, τότε αμέσως προκύπτει το ερώτημα «Έχει δουλέψει το Ινστιτούτο για αυτά τα θέματα» Σίγουρα ναι, αλλά δεν είχε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει την άποψή του. Επομένως, η μπάλα δεν βρίσκεται μόνο στο δικό σας γήπεδο, βρίσκεται και στο δικό μας. Πολύ καλά το είπατε αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Ε, να κλείσω από εδώ λέγοντα ότι πρέπει να ξέρετε ότι στη δική μα Επιτροπή έχετε, μπορείτε να βρείτε ανθρώπου που σα υποστηρίζουν. Ωστόσο, επειδή αυξάνονται οι επικρίσει και ε, πολλαπλασιάζονται τα επιχειρήματα υπέρ τη συγχώνευση των δύο αυτών Ινστιτούτων, γι' αυτό πρέπει και εμεί να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα και βασιζόμαστε σε εσά για να μα προσφέρετε λύσει για να ε, εμβαθύνουμε όλοι περισσότερο σε όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα θέματα και τελικά να καταλήξουμε να έχουμε απτά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να ε, μην δώσω το λόγο σε όλους ε, τον έχουν ζητήσει, δεν θέλω να λογοκρίνω κανέναν δηλαδή, όμως ε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Να δώσω χρόνο ε, για τρία λεπτά σε κάθε ομιλητή, διότι πρέπει και οι ομιλήτρες, οι προσκεκλημένες μας να μπορούν να απαντήσουν. Η κυρία Γκουρμάη, τρία λεπτά μόνο. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να υποδεχόμαστε και πάλι τις αξιότιμες ε, κυρίες εμπειρογνώμονες και τους συναδέλφους. Ελπίζω να περάσετε και καλά στις διακοπές. Εδώ ε, υπάρχει ένας κανόνας. Η εκπρόσωπος του ΕΛΚ μίλησε όση ώρα ήθελε. Και τώρα που ήρθε η ώρα των σοσιαλιστών με περιορίζετε και μου λέτε ότι έχω τρία λεπτά και μόνο. Δεν πάει περιπτώσει. Τι να κάνουμε ως πρόεδρος της Επιτροπής της ε, Ισότητας των Φύλων προσπαθούσα πάντα κι εγώ και οι υπόλοιποι ε, να βοηθήσω όσο μπορώ το Ινστιτούτο. Ξέραμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέξουμε τους καλύτερους εμπειρογνώμονες και είμαστε πάρα πολύ ε, περήφανοι που η δική μας Επιτροπή επέλεξε τόσο αξιόλογες ε, κυρίες για να στείλει σε αυτό το φόρουμ. Πολύ καλή επιλογή κάναμε τότε. Εκπλήσωμαι όμως λίγο. Άκουσα ότι κάνετε εκθέσεις. Πρώτη φορά τα ακούω. Γιατί δεν τις μαθαίνουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα η Επιτροπή μας. Εδώ μας έχουν λίγο αποπέδει στο Κοινοβούλιο. Επιτροπή ισότητα των φίλων και των Ευκαιριών. Μερικοί θέλουν να διαλυθούμε και τελείως, γιατί είμαστε άχρηστοι λένε. Και τώρα ακούω ότι θέλουν να καταργήσουν και το Ινστιτούτο για το Ισότητα των Φύλων. Επί μία διετία δεν συνέβη τίποτα. Ιδρύθηκε αυτό το Ινστιτούτο και στο μεταξύ χάθηκε και ο προπολογισμός Καλή η Λιθουανία και ωραία χώρα, αλλά πέφτει λίγο μακριά και γεωγραφικά και τεχνικά. Είναι δύσκολο να ε, ταξιδέψει κανείς στη Λιθουανία. Και συμφωνώ με την Edit Power, ε, θα θέλαμε να σας βλέπουμε πιο συχνά, να διαβάζουμε και τις εκθέσεις σας και να μπορούμε και να ελέγχουμε στο κάτω-κάτω ε, και τη λειτουργία και τη ποιότητα των εργασιών του Ινστιτούτου. Βεβαίως είμαι υπέρ της επικοινωνίας και είναι πολύ καλό όταν έχεις ένα προϊόν να ξέρεις και να το πουλάς εντός εισαγωγικών. Αλλά εμείς βασικά είμαστε αρμόδιοι για την ποιότητα αυτού του προϊόντος. Όχι πώς θα το πουλήσουμε, αλλά πώς παράγεται. Η ισότητα των φύλων, η ισότητα των ευκαιριών είναι κάτι που θα προαχθεί μόνο εάν κάνουμε ποιοτική δουλειά. Θα το τηρήσω το τριλεπτό κύριε Πρόεδρε, τι να κάνουμε, αλλά ε, θεωρώ επίσης ότι είναι πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας είπατε και είμαι και αισιόδοξη. Λοιπόν, αν στείλετε ξανά εκθέσεις για να φορέσετε η γραμματεία, θα φροντίσει ο Πρόεδρος να διαβιβάζονται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό ισχύει. Λυπούμε. Προσπάθησα να περιορίσω το χρόνο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας και προσπάθησα να το κάνω με όσο το δυνατόν πιο δίκαιο τρόπο. Αλλά εν πάση εκτός κάποια όρια πρέπει να κυρούνται, τηρούνται. Η κυρία Μπαραντίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τις δύο επιρρεγνώμονες για την ε, εισήγησή τους και για την εργασία που έχουν επιτελέσει, για την οποία άλλωστε διορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μία από τις ομιλήτρες μας εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ε, στη δουλειά της όντας αναπληρώτρια, διότι δεν είναι σαφή τα καθήκοντά της ανα πάσα στιγμή. Θα πρέπει σήμερα λοιπόν να επιδείξουμε ειλικρίνεια στην Επιτροπή μας και να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι οι δύο εμπειρογνώμονες είναι υπεύθυνε για όλες αυτές τις δυσκολίες που μας παρουσίασαν καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Ινστιτούτου αυτού. Επομένως, το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα η δική μας Επιτροπή έχουν εμπιστοσύνη στο Ινστιτούτο αυτό, στηρίζουν τη δουλειά του ή μήπως όχι. Αυτό είναι το ερώτημα που προκύπτει. Η Επιτροπή στηρίζει αποφασιστικά και κατηγορηματικά τη δραστηριότητα του Ινστιτούτου. Τα κράτη-μέλη στηρίζουν ε, τη δράση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου αυτού. Και αν ε, είμαστε ειλικρινεί, τότε οφείλουμε να δώσουμε αρνητική απάντηση στο ερώτημα αυτό, διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αρχή γενομένη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν είχαν πραγματική εμπιστοσύνη στο Ινστιτούτο αυτό, τότε δεν θα έθεταν υπό την ύπαρξή του, θα είχαν εδραιώσει άλλη σχέση με αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και δεν θα γινόταν καθόλου λόγο για συγχωνεύσει. Γιατί κάθε φορά βεβαίω που γίνονται περικοπέ ή πρέπει να γίνουν περικοπέ, περικοπές καλύπτονται μόνο τα πεδία που έχουν να κάνουν με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε την αυτοκριτική μας με απόλυτη ειλικρίνεια. Εμείς εδώ, εάν θέλουμε πραγματικά το Ινστιτούτο αυτό να λειτουργήσει ε, αποτελεσματικά και με επιτυχία, τότε θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει ε, πιο αποφασιστικά, ε, με περισσότερη συνοχή και συνέπεια το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και να καθορίσει τι θέλουμε εμείς αυτό να πράξει. Θέλουμε να εκτελούνται τα μέτρα ε, που υιοθετούνται από την Επιτροπή σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο. Αυτό θα ήταν καλό, κατά την άποψή μου. Θα ήταν πολύ σωστό στρατηγικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, ε, συνεπώς, είναι καλό να έχουμε καλές σχέσεις με κάθε ένα από τα κράτη-μέλη, με κάθε μία από τις ευρωπαϊκές περιφερειές και με κάθε ένα από τα Ινστιτούτα. Εγώ ε, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο πραγματικά να ε, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Και σημείο αναφοράς σημαίνει να διαθέτει τις καινοτόμες ιδέες και να συγκεντρώνει τις βέλτιστες πρακτικές που ενδεχομένως εφαρμόζονται και ισχύουν σε ορισμένες περιφέρειες, ούτω ώστε να κάνει τη διάχυση αυτών, τη διάδοση αυτών ε, στις υπόλοιπες περιφέρειες και περιοχές. Όλοι γνωρίζουμε επιτυχημένα παραδείγματα, όλοι γνωρίζουμε διαφορετικά μέτρα που ενδεχομένως έχουν επιτύχει ή όχι. Τι λείπει λοιπόν από το Ινστιτούτο. Του λείπει η στήριξη και αυτό δεν είναι πρόβλημα των εμπειρογνωμόνων οι οποίες διορίστηκαν από το κοινοβούλιο μας και αυτή τη στιγμή που ξεκινά ε, καινούρια διαδικασία δεν ξέρουν καν αν θα συνεχίσουν να κατέχουν το αξιώμα που κατέχουν. Αυτό που πρέπει εμείς να παγιώσουμε είναι η δομή ε, του Ινστιτούτου, ε, η διάρθρωσή του. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη στήριξη που του προσφέρουμε και ε, να καθορίσουμε τα συγκεκριμένα ε, μέτρα που πρέπει να ληφθούν, τα ανέφερε άλλωστε η κυρία Μανδαριάγα, ούτω ώστε να αποκτήσει νέα πνοή το Ινστιτούτο αυτό. Θα πρέπει να του χορηγήσουμε την στήριξη και σε επίπεδο προϋπολογισμού, ούτως ώστε να φέρει σε πέρα στα καθήκοντά του. Και από εκεί και πέρα να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των εργασιών του Ινστιτούτου και των δικών μας εργασιών, για να δούμε τελικά αν είμαστε διατεθειμένοι η κάθε μία και ο κάθε ένας από εμά στο βαθμό που εκπροσωπούμε συγκεκριμένο κράτος ή συγκεκριμένη περιφέρεια, τελικά τα μέτρα που, παρουσιάζει το Ινστιτούτο να διαδοθούν ε, στην περιοχή μας ή στο κράτος μας ώστε ε, να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές παντού. Ε, θέλω να ευχαριστήσω τις ομιλήτριες και να επιμείνω στο ότι εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά που μας αναλογεί, πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Είναι εύκολο να δοθεί νέα πνοή στην ε, λειτουργία του Ινστιτούτου. Το μόνο που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση, η οποία με πάσα ειλικρίνεια απουσιάζει κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ η κυρία Λιωτάχ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω ε, και τα δύο μέλη ε, για τη σαφή ε, παρουσίαση που μας έκανα και των θετικών και των αρνητικών ή των πιο συζητήσιμων σημείων. Γιατί όταν αναφέρουμε τα σημεία κριτικής μπορούμε να προχωρήσουμε. Για το Ινστιτούτο νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει πολύτιμη συνεισφορά εάν, λειτουργεί, και εάν λειτουργήσει τελικά σωστά. Έχω μια ερώτηση και προς ε, τα δύο μέλη. Μας ανέφεραν τα πιο κρίσιμα σημεία, σημεία που επιδέχονται κριτική. Τα έχετε συζητήσει και με τα μέλη του Ινστιτούτου. Έχετε μια λίστα, έχετε ένα κατάλογο που θέλετε να συζητήσετε και μαζί μας. Ε, έχω σημειώσει και τα θέματα της επικοινωνίας που αναφέρετε ε, και μεταξύ ημών με ύψιλον και ημών με ήτα. Αυτό εύκολα μπορεί να λυθεί και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Πρόεδρο σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις των συντονιστών να συμφωνήσουμε και να καταλήξουμε για το πώς θα επικοινωνούμε. Ε, καλύτερα με ε, τους εμπειρογνώμονες και με το Ινστιτούτο και να κοιτάξουμε γιατί συνέβη αυτό. Το είπε και η κυρία Μπάουερ. Όταν ζητούμε και αναθέτουμε εκθέσεις και τα λοιπά, γιατί δεν το κάνουμε μέσω του Ινστιτούτου. Γιατί τα αναθέτουμε σε εξωτερικούς. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες, ειδικοί λόγοι. Ε, για να το συζητήσουμε. Και για τις ακροάσεις. Καλό θα ήταν να καλούμε εκεί εμπειρογνώμονες, ειδικού, αν μη τι άλλο να είναι παρόντες για να υπάρχει μια καλύτερη σύνδεση και με τον πολιτικό κόσμο και τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα που εμείς συζητούμε. Αν θέλουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το Ινστιτούτο, θα πρέπει και εκείνοι να ξέρουν τι θέματα μας απασχολούν καθημερινά στην Επιτροπή μας. Να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε, αλλά να έχουμε και συγκεκριμένες προτάσεις αλλά από μέσα, ε, από το ίδιο το Ινστιτούτο, πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στις ε, προσκεκλημένες μας. Παρακαλώ, για το λόγο να απαντήσετε στα ερωτήματα που ετέθησαν και στα σχόλια, αν το επιθυμείτε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. διαπιστώνω ότι έχουμε τα ίδια μελήματα και τις ίδιες ανησυχίες. Τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, μπορούν να πάνε καλύτερα και πρέπει να πάνε καλύτερα. Θα ήθελα να σας πω ποιο προβλέπω ως πρόβλημα ε, και να το μοιραστώ μαζί σας. Όλα αυτά τα κάνουμε εμείς στον ελεύθερο χρόνο μας. Ούτε πληρωνόμαστε ε, και επίσης και τα ταξίδια Ας πούμε εγώ την ώρα που είμαι εδώ στην Επιτροπή δεν μπορώ να κερδίσω χρήματα από άλλη δραστηριότητα και αυτό είναι πρόβλημα και θέλω να το πω. Στη συνέχεια, ε, κατάλογο συστάσεων λέτε. Θα σας τα διαβιβάσουμε, μπορούμε να τα, σας, στείλουμε με mail, δεν χρειάζεται να είμαστε ε, ε στη διέθουσα και μέσα σε 1,5-2 μήνες ε, μπορώ να σας έχω στείλει ένα κατάλογο με συστάσεις και προς εσάς αλλά και στο ίδιο το Ινστιτούτο. Πουθενά δεν έχουμε καμία εξουσία εμείς, ούτε σε εσά ούτε στο Ινστιτούτο. Θα πρέπει να βασιστούμε στη δύναμη της πυθούς μας. Ε, μία σύσταση, για παράδειγμα, θα ήταν να πούμε στο Ινστιτούτο ότι όταν κάνετε προσλήψεις να τους στείλετε για στάζ, άσκηση, είτε στο Κοινοβούλιο, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια εβδομάδα στο κάθε όργανο και μερικές μέρες και στο Συμβούλιο, για να γνωρίζουν τα θέματα από πρώτο χέρι. Τέτοιες συστάσεις μπορούμε να τις κάνουμε. Ε, και ελπίζω να εισακουστούν σε σχέση με τα όσα είπε η κυρία Λιωτάρ. Γιατί το Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει διάφορες μελέτες και έρευνες σε τρίτους και όχι στα δικά μας όργανα, δεν το γνωρίζω. Ε, θα έχουν τους λόγους τους. Αλλά ξέρω ότι και στο Ινστιτούτο γίνονται μελέτες τις οποίες αναθέτουν και αυτοί σε τρίτους στους ίδιους που τις αναθέτετε και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται λοιπόν συντονισμός να μην γίνονται τρεις εκθέσεις για το ίδιο θέμα. Ε, δηλαδή μια φορά σε εσά, μια φορά στην Κομισιόν και μια φορά στο Ινστιτούτο. Κρίμα, είναι πεταμένα λεφτά. Για τη στρατηγική επικοινωνίας, ε, το σημειώνω με χαρά. Και το θέμα της πολιτικής βούλησης για τη συγχώνευση δεν το θίγω, γι' αυτό το αφήνω στην άκρη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Bueno, eh, Λοιπόν, ε, είναι προφανές ότι δεν θα θίξω τα ίδια θέματα με την συνάδελφο, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου, μεγαλύτερη ανησυχία με αυτή από ό,τι ήλθα. Ε, εγώ ήρθα εδώ για να ζητήσω εμπιστοσύνη προς το Ινστιτούτο και συνεργασία από τους ευρωπαϊκούς ασμικούς φορείς προς το Ινστιτούτο και τι βλέπω τελικά ότι με την ε, συγχώνευση που τελικά προτείνεται, προτείνεται με το άλλο Ινστιτούτο, με τον άλλο φορέα, να καταστεί πραγματικά τελείως ανύπαρκτη ε, η ύπαρξή του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή είναι άγνωστο και δεν είναι σημείο αναφοράς και θέλουμε να γίνει σημείο αναφοράς, το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί είναι να συγχωνευτεί με έναν άλλο φορέα, γιατί τότε είναι που θα εξαφανιστεί εντελώς. Πιστεύω ότι πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό το ζήτημα και με όλους όσους το θέτουν στο τραπέζι. Τι μπορούμε να κάνουμε όλες μας για να το βελτιώσουμε το Ινστιτούτο, να του δώσουμε μια νέα όθηση, να το λανσάρουμε εκ νέου, ναι. Όλα είναι πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε. Όμως όλα αυτά δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα αν ταυτόχρονα συγχωνευτεί α, και ουσιαστικά εξαφανιστεί από έναν άλλον οργανισμό. Όπως πολύ ορθά είπε συνάδελφος Βίλεμ, με χαρά να σας υποβάλουμε προτάσεις υπό τη μορφή συστάσεων, αλλά θα θέλαμε και εμείς από πλευράς μας να ακούσουμε ποια είναι η δική σας άποψη και ιδίως η άποψη της δικής σας επιτροπή για το μέλλον του Ινστιτούτου. Αν τελικά και εσείς βλέπετε το μέλλον του είναι συγχώνευση με κάποιον άλλο φορέα, τότε δεν έχει νόημα όλο αυτό και θα πάει και στράφει όλο το έργο που έχει γίνει. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ευαισθητοποίηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες και αυτό αφορά όλους τους ευρωπαϊκούς εθνικούς περιφερειακούς φορείς που ασχολούνται με θέματα ισότητας των φύλων. Κάθε Ινστιτούτο χρειάζεται μία ενίσχυση, μία βοήθεια για να αποτελέσει σημείο αναφοράς, για να α, έχει ένα εκτόπισμα, να έχει μια σημασία, Χρειάζεται λοιπόν μια ενίσχυση. Η συγχώνευση είναι το αντίθετο. Είναι σαν να είναι μια ψυχρολουσία, ε, αν θέλετε, και φέρνει τα τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Με ανησυχεί λοιπόν τα μάλα αυτή η πρόταση. Γιατί φαίνεται ότι είναι μια πρόταση που είναι στο τραπέζι τελικά, στο τραπέζι εργασίας και αποτελεί μια δυνατότητα τελικά. Εμείς πιστεύουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία στο Ινστιτούτο με τη βοήθεια όλων. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να εμπιστευόμαστε πρώτα απ' όλα τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο. Άρα και αφήστε τη στιγμή στο Ινστιτούτο το παιδί που έφερε στον κόσμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το επιδείξετε μια κάποια α, εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να το βοηθήσετε, να το στηρίξετε και να του ξεκαθαρίσετε τον ρόλο που πρέπει να έχει αυτό το Ινστιτούτο και για να μπορέσει να αποτελέσει μια αναφορά σε σχέση με όλους τους συναφείς φορείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η δική μου θέση ως εμπειρογνώμονας και ως ε, συμμετέχουσα στο φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Αν το κάνετε αυτό, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευράς μας, κάθε προσπάθεια για να προχωρήσει το Ινστιτούτο να αποτελεί σημείο αναφοράς. Αλλά ταυτόχρονα, επαναλαμβάνω, χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό όλοι όσοι δουλεύουν στο Ινστιτούτο θέλουν κάποιε προποθέσει, κάποια εχέγγυα. γιατί, επαναλαμβάνω, εμείς δεν εργαζόμεθα στο Ινστιτούτο ε, επαμοιβή, δεν εργαζόμαστε εκεί καθημερινά, δεν είναι η κυρία μας απασχόληση. Για να μπορέσουμε λοιπόν να το βοηθήσουμε και τον ενισχύσουμε, χρειάζεται μία επιπρόσθετη προσπάθεια από όλους μας. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να στηρίξουμε, να βάλουμε πλάτη για να μπορέσει να προχωρήσει ε, και να επιβιώσει το αυτό. Είναι λοιπόν το αίτημα που απευθύνω σε εσά. Να επανέλθουμε εδώ και να συζητήσουμε το μέλλον του Ινστιτούτου και να αφήσουμε το θέμα στην άκρη. Βεβαίω από εκεί πέρα εμεί σεβόμεθα τη δική σα θέση και εσεί θα αποφασίσετε. Eh, Ευχαριστούμε πολύ. Θα προσπαθήσω και εγώ από πλευρά μου να διατρέξω κάποια ζητήματα, να πω ότι η Επιτροπή αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει επιδείξει ήδη την απόλυτη εμπιστοσύνη της προς το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και θέλουμε να συνεχίσει ε, να ε, υπάρχει και να δίνει έργο. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετά γνωστό. Ε, δεν υπάρχει προβολή και ορατότητα του έργου του Ινστιτούτου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν, ως σύνολο, όχι μόνο η Επιτροπή μας, θα ξαναδεί το θέμα της συγχώνευσης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου με το FRA. Α, έως σήμερα η Επιτροπή μας δεν έχει υποστηρίξει αυτή τη θέση συγχώνευσης, όμως είναι δύσκολο να ανατρέψουμε αυτή την τάση που υπάρχει στο Παγκοκοινοβούλιο. Ήδη δεν υπάρχει μια απόφαση, δεν, έχει, ε, κάποια, δεν είχε ληφθεί κάποια απόφαση, υπάρχει μια τάση. Ε, είναι λοιπόν ευθύνη όλων μας αυτή τη στιγμή εφόσον υποστηρίζουμε ε, το Ινστιτούτο ως ε, παρουσία αυθύπαρκτη, να το στηρίξουμε ώστε να δώσει αποτελέσματα και έργο. Συμφωνώ λοιπόν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά να μην παραγνωρίσουμε ότι γίνεται και η συζήτηση για τη συγχώνευση. Πιστεύω ότι όσοι πήραν το λόγο ήταν ξεκάθαροι στι θέσει του και έκαναν πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Ακούστηκαν και πολύ ενδιαφέρουσε προτάσει τι οποίε μπορούμε να επεξεργαστούμε στο μέλλον. Ακούστηκαν ε, προτάσει όπω ένα κατάλογο κατάλογος συστάσεων. Ήταν μια εξαιρετική πρόταση. Και αυτό που είπε η κυρία Λωτά ήταν, πιστεύω, εξίσου εύστοχο να το δούμε τη συνεδρία των συντονιστών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να γίνει στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών αυτό, αλλά τουλάχιστον σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις των ιστών θα συζητηθεί για αυτό το θέμα. Θέλω και πάλι να ευχαριστώ θερμά τις προκεκλημένες μας για τον χρόνο που μας αφιέρωσαν. Ήταν πραγματικά πολύτιμη αυτή η συζήτηση. Και ήταν πραγματικά εξαιρετικό που ταξιδέψατε ε, για να έρθετε μέχρι εδώ, για να ανταλλάξετε απόψεις μαζί μας. Ήταν μια επικοδομητική τελεγή απόψεων, γιατί ακούστηκαν πολύ εύστοκες προτάσεις. Ευχαριστώ όλους θερμά. Καλώς. Προχωρούμε λοιπόν στην υπερήσια διάταξη. Είμαστε στο σημείο 10, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Εφαρμογή των προτεραιοτήτων για το 2012.